Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. Άρχεται η συνεδρίαση. Vous avez vu le projet d'agenda. Euh, έχετε λάβει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, το έχετε κοιτάξει. Εάν δεν έχετε σχόλια, θεωρείτε εγκριθεί σε ημερήσια διάταξη. Γύρω στις 4.30 έχουμε προβλέψει ώρα ψηφοφορίας για μία ώρα. Το λέγω και για τα παράοντα μέλη, αλλά και για τα απόντα. Για να τους το διαβιβάσουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ομάδων, έτσι ώστε να έχουμε αρκετά μέλη για να ψηφίσουμε. Ε, παρτία δηλαδή. Je vous, ε, ε, Θα σας πρότεινα να προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη ε, κάτι, όχι ξεχωριστό θέμα, στο 4 να εντάξουμε ένα ζήτημα που είναι το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 2013 για την ένταξη της Κροατίας. Πριν από λίγες μέρες κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον τριμερή διάλογο αναφερθήκαμε λίγο σε αυτό επιγραμματικά. Ο ζήτη για το 2014, 2013, συγγνώμη, ε, αν παρευρίσκεται θα μπορούσε να μας ενημερώσει σχετικά. Αυτά. Το θέμα για τα κτίρια Πρέπει να σας πω ότι η μόνιμη συγκήτριά μας, η κυρία Χολμαϊέρ, απουσιάζει και ζητεί συγγνώμη, είναι δικαιολογημένους απούσα, αλλά ανέθεσε στην κυρία Σουζάνα Πόρσο που είναι από άλλη πολιτική ομάδα βέβαια, αλλά με την οποία συνεργάζεται mm. ε, απρόσκοπτα να μας παρουσιάσει το θέμα. Βέβαια η Σουζάνα δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ανακοινώσεις του Προέδρου θα το βρείτε στο Κόμπου News ή Buds Newsletter, όπως λέγεται τώρα και θα πρότεινα να έρθουμε αμέσως στον προπολογισμό του 2014 πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων. Δίναμε στο λόγο στην εισηγήτριά μας, Αν Ιένσεν. Yes, thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου Και από τότε προχωρήσαμε λιγάκι στη συζήτηση των ημερομηνιών του χρονοδιαγράμματος τη συνέχεια του τριμερούς διαλόγου τον Ιούλιο και το λέει το αυτό στα νέα της κομπούς. Προς στιγμήν επισκέπτομαι τις επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές για να περιγράψω την κατάσταση και να ξέρουν και αυτοί να μας πούνε πώς βλέπουν τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων. <clears throat> και διαπίστωσα ότι όλες οι επιτροπές έχουν συγκεκριμένες ιδέες για το και ως προς τις δυσκολίες στο νομικό υπόβαθρο που δεν υπάρχει το Πολδίπ, αλλά επίσης οι επιτροπές συνεχίζουν να συζητούν ιδίω στην νομοθετική βάση και οι περισσότερες έχουν ξεκάθαρισμένες ιδέες ως προς την κατεύθυνση που θέλουν να πάρει ο προϋπολογισμός. Δεν φοβάμαι λοιπόν καθόλου μήπως εμείς το Κοινοβούλιο δεν καταφέρουμε να έχουμε σαφή θέση επί του προϋπολογισμού παρά τη δύσκολη φάση που αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε ακόμη οριστική ημερομηνία από την Κομισιόν για το πότε θα υποβάλει τον προϋπολογισμό. Μέσα Μαΐου έχει πει, αλλά επίσης είπε τέλη Μαΐου. Και φαντάζομαι ότι τα τέλη Μαΐου προτιμούν τελικά. Και άρα μάλλον θα πιεστούν οι συγκεκριμένοι μεμονωμένες επιτροπές και οι δικοί μας μέχρι να καταλήξουν σε συγκεκριμένη εντολή για τον Ιούλιο. Αλλά, όπως γράφει και εδώ, είναι δυνατόν στις 19 Ιουνίου να γίνει ανταλλαγή απόψεων ενός σχεδίου προϋπολογισμού και άρα θα έχουμε τρεις εβδομάδες για να αν είναι τέλη Μαΐου δηλαδή που θα το υποβάλουν για να φτάσουμε μέχρι την 21η Ιουνίου που είναι η διορία υποβολής των χρονοδοτήσεων των μεμονωμένων επιτροπών. Μετά θα οριστεί η προθεσμία των τροπολογιών και αυτή η 21η Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Όπως βλέπετε λοιπόν είναι πολύ πιεστικό το χρονοδιάγραμμα και μάλλον αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταφέρουμε πολλά ακατόρθωτα πράγματα όπως τις πλήρεις μεταφράσεις και ε, δεν μπορούμε μόνο με τα αγγλικά να τα καταφέρουμε αλλά θα το προσπαθήσουμε για να ετοιμάσουμε λοιπόν τον τριμερή διάλογο του Ιουλίου και να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι χρήσιμο για να έχει κάποιο νόημα ο διάλογος αυτός. Αυτά είχα να σας πω βασικά. Ευχαριστούμε Άννα. Φέτος όντως, λόγω της καθυστέρησης του Συμβουλίου στην εξέταση του Πολβίπ, οι διαπραγματεύσεις του τώρα θα αρχίσουν και η Κομισιόν είναι σε δύσκολη θέση γιατί δεν ξέρει σε ποια ακριβώς βάση να προετοιμάσει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014 που φυσικά πρέπει να ακολουθεί τα ανώτατα όρια που θα ορίσει το Πολδίπ. Ήδη την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε το θέμα και ενθαρρύναμε την Κομισιόν να βασιστεί στις αρχικές προτάσεις που μας είχε κάνει στο σχέδιο Πολδίπ. Εν τω μεταξύ όμως το Συμβούλιο έλαβε διαφορετική θέση για τους αριθμούς και την ανώτατα όρια, τις οροφές και γι' αυτό με την ευκαιρία του διαλόγου της προηγούμενης εβδομάδας και τη συζήτησή μας με τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι είχα πει ότι η ευθύνη της Κομισιόν είναι να καθορίσει τους ακριβείς αριθμούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις τεχνικές δυνατότητες που έχουμε απορρόφησης και στις πολιτικές δυνατότητες επίτευξης συμφωνίας. Αυτή είναι η ευθύνη της Κομισιόν. Και επέμεινα επίσης να τηρήσει ένα χρονοδιάγραμμα η Κομισιόν τέτοιο που να επιτρέπει και στις δύο πλευρές της αρχής του προλογισμού, δηλαδή και του Κοινοβούλιο, επαρκή χρόνο για να μπορέσουν να το επεξεργαστούν και τελικά οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να μπορέσουν να υποβάλουν και τροπολογίες. Η Επιτροπή Προπολογισμών επίσης να καταθέσει και να εγκρίνει τροπολογίες και οι πολιτικές ομάδες να έχουν επαρκή χρόνο μέχρι την Ολομέλεια για να τα επεξεργαστούν και εκείνες. Όπως είπε και η Άννα λοιπόν, η Κομισιόν βασίζεται μάλλον στην υπόθεση έγκρισης από την Κομισιόν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Την Τετάρτη εκείνης της τελευταίας εβδομάδας, 29, προβλέπουμε την επομένη να έχουμε ολόκληρη μέρα συνεδρίαση για να δούμε αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε ή να κάνουμε μισή μέρα νωρίτερα τη συνεδρίαση της Κομπούς ώστε σύμφωνα με τα Ιωθώτα επί των οποίων θέλω να επιμείνω, ο Επίτροπος Αρμόδιος για τον Προπολογισμό να έρθει να μας παρουσιάσει στην Επιτροπή μας τη θέση της Κομισιόν πριν τη σχολιάσει τον τύπο. Παράλληλα, η Κομισιόν ενέκρινε ένα σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 13 για την ένταξη της Κροατία. της Κροατίας τα πράγματα προχωρούν όπως είχαν προβλεφθεί και δεν φαίνεται να τεθεί καμιά δυσκολία για την θέση ενισχύ 1η Ιουλίου της ενταξιακής αυτής συνθήκης. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει λοιπόν και πρέπει τώρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ο διορθωτικός προϋπολογισμός να εγκριθεί εν ώστε να εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και στην Κροατία. Μάθαμε δε σήμερα ότι αύριο η Κομισιόν θα υποβάλει τον διορθωτικό προπολογισμό 2 που θα επιτρέψει πρόσθετα κοντήλια για την Ένωση και για να εφαρμόσει δεσμεύσεις που είχε αναλάβει και που δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί και για να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες του 13 όπως έχουν προβλεφθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα. Για το διορθωτικό προπολογισμό του 13 λοιπόν ο Τζοβάνι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως έλεγες, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου από την Επιτροπή. Ο στόχος του είναι να συμπεριλάβει στον προπολογισμό του 2013 τα αναγκαία ποσά σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και τις πληρωμές για την κάλυψη των ε, δαπανών που είναι συναφής με την ένταξη της Κροατίας ως 28ο έτος της Ένωσης από την 1η Ιουλίου του 2013 και μετά. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο καλύπτει τις δαπάνες για την Κροατία για τα επόμενα 7 χρόνια. Τούτο είναι αναγκαίο για το 2013 για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δαπάνες για το τελευταίο εξάμεινο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα με το πρώτο διορθωτικό προπολογισμό του 2013 η Επιτροπή υπέβαλε και πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου για να το τροποποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης όπως βλέπετε από το άρθρο 29 της ε, Διοργανικής Συμφωνίας. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός παριθμών 1 προβλέπει αύξηση 556 εκατομμυρίων ευρώ σε δεσμεύσεις και 374 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμές. Κάτι που ευθυγραμμίζεται με αυτό που προβλέπει η Συμφωνία Προσχώρησης και που καλύπτουν μόνο τις λειτουργικές δαπάνες, δεδομένου ότι οι διοικητικέ δαπάνε ε, τη κατηγορία 5 ήδη συμπεριλαμβάνονται στον προπολογισμό του 2013. Είχαμε ήδη δηλώσει ότι δεν θα προβλέπαμε καμία αλλαγή στον προπολογισμό για να λάβουμε υπόψη την είσοδο στην Ένωση της Κροατίας. Στον φετινό πρώτο τρίλογο που έγινε 19 Μαρτίου και αυτός υποβάλαμε στο Συμβούλιο μαζί με την αντιπροσωπεία που εκπροσωπούσε το Κοινοβούλιο την ε, τεχνική και όχι πολιτική διάσταση αυτού του διορθωτικού προπολογισμού. Και μάλιστα παρά τις προβλέψεις αναθεώρησης των ανωτάτων ε, όδιων για το πολιετές μεσονομικό πλαίσιο του 2013 που οφείλεται στην εφαρμογή των όσων προβλέπονται μέσω της διοργανικής συμφωνίας και στην ε, συμφωνία ένταξης, ζήτησα ο προϋπολογισμός, ο διαφορετικός αυτός προϋπολογισμός να γίνει με μια μικρή τεχνική αλλαγή που θα λάβει υπόψη την πολιτική συζήτηση μετά, τις ε, διαδοχικ... μετά τους διαδοχικούς προϋπολογισμούς, για να καλύψουν τις ε, πληρωμές των Ρέστα ε, Λικιντέ του 2012. Αύριο θα υπάρξει έγκριση του δεύτερου διορθωτικού προπολογισμού από πλευρά τη Επιτροπή. Με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου τονίσαμε στον τρίλογο ότι για το Κοινοβούλιο η μόνη δυνατότητα πληρωμών στον ε, διευθυντικό προϋπολογισμό είναι της προσφυγής στους νέους και πρόσθετους πόρους, αποφεύγοντας δηλαδή οποιαδήποτε, οποιοδήποτε ενδεχόμενο reading blocking, σε ό,τι αφορά το χρονικό ορίζοντα για την εξέταση του προϋπολογισμού υπαριθμών 1 ζητήσαμε να επιταχύνει τη διαδικασία έγκριση στο Συμβούλιο και να μην περιμένουμε ολόκληρες 8 εβδομάδες που προβλέπονται από τα εθνικά κοινό, για την ε, άποψη των εθνικών κοινοβουλίων για να έχουμε χρήσιμο χρόνο ούτως ώστε να έχουμε εγκρίνει το κείμενο αυτό μέχρι την 1η εβδόμου του 2013 οπότε θα γίνει πλήρες μέλος της Ένωση η Κροατία. Από πλευρά του το Συμβούλιο δήλωσε ότι θα ξεκινήσει ε, τη σχετική εξέταση. Εμεί περιμένουμε τη θέση του Συμβουλίου και θα αναλάβουμε την απαραίτητη δράση κατόπιν. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να αναμένει τις 8 εβδομάδες, το χρονοδιάγραμμά μας θα επιταχυνθεί. Μπορεί να προβλέψουμε ψηφοφορία στις 8, στις 7 Μαΐου, πριν την τελική ημερομηνία του ψηφοφορία στο Συμβούλιο, ή 16-30 Μαΐου, μετά την ε, ψηφοφορία και ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ιουνίου που είναι η μόνη προθεσμία που μπορούμε να τηρήσουμε για να έχουμε την έγκριση του προπολογισμού, του διευθυντικού προπολογισμού πριν την επίσημη προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση. Το σχέδιο έκθεσης μπορεί να υποβληθεί είτε στις 24-25 Απριλίου με προθεσμία για τις τροπολογίες πάνω κάτω ανάλογα με την ημερομηνία που θα επιλέξουμε για την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω εκ νέου είναι ότι ο διορθωτικός αυτός προϋπολογισμός έχει καθαρά τεχνική φύση για να προσαρμόσει τις δεσμεύσεις και τις πληρωμές και τα μέγιστα όρια των ε, ε πολιετών, ε, του πολιετού μεσονομικού πλαισίου στις νέες συνθήκες μετά την ε, ένταξη της Κροατίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι μόνο η... σε αυτό το πλαίσιο μόνο νέοι πόροι μπορεί να ληφθούν υπόψη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Τζοβάνι. Ο Σαλβαντόρ. Και αυτό θέλω και εγώ να ρωτήσω τον Τζοβάνι. Ας υποθέσουμε ότι το Συμβούλιο θα μιλήσει για αναδιάταξη ε, των γραμμών και ε, όχι αλλαγή των ανωτάτων ορίων. Εμείς ως Κοινοβούλιο τι θα επιλέξουμε, μια ενδιάμεση λύση γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του Συμβουλίου. Μα μιλούμε για το προϋπολογισμό της Κροατίας, έτσι δεν είναι. Όχι για το, τους εκτάκτους διορθωτικούς προϋπολογισμούς για το 2013. Εμείς ως πολιτική προτεραιότητα και μοναδική δυνατότητα έχουμε το διορθωτικό προϋπολογισμό για την Κροατία και να έχει αποκλειστικά νέους πόρους. Αυτό όμως χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Υπάρχει εκεί κανένα περιοθώριο διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο ή για μας είναι ένα θέμα αποκλειστικά τεχνικό όπως λέγει ο εισηγητής. Οπότε δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Εν περιπτώσει. Η αντίδραση του Συμβουλίου για το διαρθρωτικό προϋπολογισμό για την Κροατία θα μας δείξει και τη γενικότερη στάση του για άλλους προϋπολογισμούς διαρθρωτικούς ε, με υψηλότερα ποσά από αυτά της Κροατίας. Merci Salvador. Giovanni. Giovanni. Κοιτάξτε, η προσέγγιση που είχαμε στον τρίλογο να υποβάλουμε δηλαδή την πρόταση αυτή ως έναν τεχνικού χαρακτήρα διορθωτικό προϋπολογισμό που συνδέεται με την ε, συνθήκη προσχώρησης για να λάβουμε υπόψη βεβαίως στην ε, φύση του διορθωτικού προϋπολογισμού μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να σας πω ότι σε μια χρήση το 2013 όπου οι πληρωμές Ξέρουμε ότι είναι ανεπαρκής, όλοι το ξέρουμε ότι δεν μπορούν να καλύψουν και τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Το να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το redeployment για να καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από την άφηξη ενό νέου κράτου μέλους δεν είναι εύκολα κατανοητό. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Συμβούλιο πρέπει να δείξει μια ισχυρή ε, πολιτική βούληση και δεν μιλάμε και για μεγάλα νούμερα στις πληρωμές ε, το ποσό που μιλάμε είναι της τάξης ε, των 374 εκατομμυρίων ευρώ. Το να επαναφέρουμε το redeployment, τη μεταφορά δηλαδή από μία κατηγορία σε άλλη, έχει μια ισχυρή είναι ένα τεχνικό εργαλείο που αμφισβητεί την πολιτική σημασία της διεύρυνσης. Και νομίζω ότι το, είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει νέους πόρους στο Συμβούλιο, μεταξύ άλλων και διότι αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε ή να θέτουμε υποσυζήτηση για το πλαίσιο του redeployment, τις πιθανές κρίσεις στο Συμβούλιο ως προς τον διορθωτικό προϋπολογισμό που αύριο θα έπρεπε να εγκρίνει η Επιτροπή στο Κολέγιο των Επιτρόπων και που θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες τι θα σίγουρα θα αφορά ποσότητες αρκετά υψηλότερες, ποσά αρκετά υψηλότερα. Ευχαριστώ. Έχω μπροστά μου τις διατάξεις της βιστάμενης διοργανικής συμφωνίας. Παράγραφος 29. Αν νέα κρατημέλη προσχωρήσουν στην Ένωση κατά τη διάρκεια της περίοδου που καλύπτεται από το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με το σημείο 3, από κοινού θα αντιμετωπίσουν θα αλλάξουν το δημοσιονομικό πλαίσιο για να λάβουν υπόψη τις απαραίτητε δαπάνε που προκύπτουν από την έκβαση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Είναι σαφές για έναν κανονικό αναγνώστη, όχι για έναν Υπουργό Οικονομικών αναγκαστικά. Σίγουρα λοιπόν θα έχουν μια συζήτηση μεταξύ τους. Η πρόταση της Επιτροπής μου φαίνεται εύλογη. Λέει ότι οι διοικητικές δαπάνες κάπως τα βγάζουμε πέρα αλλά για τις επιχειρησιακές λειτουργικές ανάγκες, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της παραγράφου 29, είναι λογικό να υπάρξει προσαρμογή των των ορίων. Θα δούμε. Θα με εξέπλητε αν δημιουργούσε δυσκολίες στο Συμβούλιο, που θα είχαν επίπτωση την καθυστέρηση μιας συμφωνίας που δεν θα δείχνει ότι το νέο, μέτρος, μέλος, η Κροατία δηλαδή, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Βεβαίως, βλέποντας το πώς αντιμετώπισε την Κύπρο το Συμβούλιο, θα έλεγα ότι όλα είναι δυνατά αν μπορούμε να τσακίσουμε τα μικρά κράτη της Ένωσης. Θα δούμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Αύριο με ενημέρωσε, ο κ. Ζεβαντόφσκι με ενημέρωσε, μάλλον ο κ. Ζεβαντόφσκι με ενημέρωσε επίσημα ότι αύριο η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ε, υπαριθμό 2 διορθωτικό προπολογισμό. με τον όρο που περιγράφει ως Big Bang. Ο κ. Λεβαντόφσκι ήταν έτοιμος να έρθει στους, είναι έτοιμος να έρθει αύριο το απόγευμα στους συντονιστές μιλήσαμε στο τηλέφωνο τώρα το απόγευμα, τον ευχαρίστησα, αλλά για πρακτικούς λόγους δεν θεωρήθηκε ότι τούτο είναι σωστή, δεδειγμένη λύση. Συμφωνήσαμε μαζί του να οργανώσουμε μία έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Προπολογισμών τη Δευτέρα το βράδυ του επόμενου Στρασβούργου για να μπορέσει να έρθει ο Επίτροπος να μας παρουσιάσει το Big Bang με λεπτομέρεια και μετά ο εισηγητής και όλοι σας θα μπορείτε να θέσετε όλα τα ερωτήματα που θεωρείτε σκόπιμα στον Επίτροπο. Η σχέση μεταξύ της επίλυσης του προβλήματος των πληρωμών του 2013 και των διαπραγματεύσεων ε, για το MFF 2014-2020 περιλαμβάνεται στο ψήφισμα που υιοθετήσαμε στις 13 Μαρτίου με μεγάλη πλειοψηφία. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευρά μα τουλάχιστον, ούτω ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσει στην εξέλιξη των διαφόρων προτάσεων. Ω προ την εκτέλεση 2013-2014 δεν βλέπω άλλε παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή. πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Δεν βλέπω να θέλουν να μιλήσουν οι συγγητές. Κανείς άλλος δεν θέλει το λόγο. Ωραία. Τόσο πολύ που το συζητάμε, προφανώς δεν χρειάζεται να το συζητάμε πάντα. Τώρα προτείνω. Ήρθε η κυρία Μποζομποράτα. Από ό,τι βλέπω η κυρία Χολμάγερ σας ζήτησε να μιλήσετε για το σημείο 14 που είναι το δικό της θέμα, την πολιτική ακινήτων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα εξ ονόματος ε, της Μόνικα Χολμάγερ να σας ενημερώσω. Με παρακάλεσε να αναλάβω αυτό το θέμα για το μεταφραστικό κέντρο στο Λουξεμβούργο. Είναι δύο τα κτίρια τα οποία μισώνουμε και προσεχώς θα μετακινηθούν σε ένα κτίριο, το οποίο ε, έχει μετασκευαστεί, έχουν γίνει διάφορες εργασίες, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Ε, στις 15 Απριλίου αποφασίστηκε να τερματιστεί η μίσθωση του ενός κτηρίου 1,86 εκατομμύρια ετησίως ήταν το μίσθωμα, ε, λίγο πιο ακριβό από αυτό που καταβάλλεται τώρα. Ε, υπάρχει δυνατότητα μείωσης κάπως περιστολής του κόστους καταφέραμε κάπως να το περιορίσουμε, η διαφορά μπορεί να μην ήταν πολύ μεγάλη, ε, Παρ' αυτά καταφέραμε να κάνουμε κάποιες οικονομίες. Ε, γίνονται και άλλες διαπραγματεύσεις. Ας πούμε, για ένα δίμηνο δεν θα πληρώσουμε καθόλου ενίκιο και ε, το κτίριο ανήκει στο κράτος του Λουξεμβούργου ζητούσαν ετησίως ε, ένα μίσθωμα της τάξης των 240.000 Το μεταφραστικό κέντρο αυτό προσπαθώντα να δούμε πόσο ο χρηματοοικονομικός κανονισμός μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό. Δεδομένων λοιπόν των δυσκολιών και των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην ΑΦΚΟ, μπορούμε να το δουλέψουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να ετοιμάσουμε τροπολογίε και να μπορέσει η συγκίτρια μας να βρει συμβιβαστικέ ε, προτάσεις. Η προθεσμία λοιπόν για την έκθεση της ΙΝΚΕ μετατίθεται για τις 29 Απριλίου ώρα 12. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Προτείνω να πάμε στο σημείο 7. Έκθεση Ταχντέν που μόλις ε, είδα ότι φτάνει, αλλά δεν ξέρω που είναι. Να τους. Πολύ αριστερά σήμερα. Για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση προ όφελο τη Αυστρία για ένα αυστριακό έργο. Κύριε Σιγητά, Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω. Θα μιλήσω μόνο για τους απολυμμένους εργαζόμενους, τους 270, για τους οποίους ζητιέται ένα ποσό εδώ από την Αυστρία, και το ποσό αυτό καλύπτει διάφορες δραστηριότητες που προτείνεται να αναλάβουν Έχω καταθέσει μερικές τροπολογίες που ανταποκρίνονται ακριβώς στην επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης προς τη δική μας και σας πληροφορώ ότι την τελευταία, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης είχαμε πει να θέσουμε το θέμα στον τριμερή διάλογο για τη διαχείριση δηλαδή του Ταμείου Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστούμε. ένα σχόλιο. Όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για το θέμα αυτό θα ψηφίσουμε στις, σε λίγα λεπτά σήμερα. Στις 26 Μαρτίου έγραφε. Το ίδιο και για το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Η συγγήτρια του 7 δεν ήταν παρούσα, του 6 μάλλον η Αγγέλικα Βέρτμαν, αλλά μπορούμε, μήπως ο κύριος Νταρντένο εισηγητής του 7 έχει να μας πει τίποτα, όχι. Ναι, πρόκειται για τις ε, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και 3,7 εκατομμύρια προβλέπονται. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο πρόσφατες περιπτώσεις που δείχνουν πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το ταμείο και Ξέρετε ότι από αυτού υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και στο Συμβούλιο και μέσα στο Κοινοβούλιο για τη διαπραγμάτευση του επόμενου πολιτικού. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλά τα είπαμε μέχρι τώρα. Χειριστήκαμε πολλά θέματα, αυτά που προβλεπόταν δηλαδή πριν την ψηφοφορία. Στρέφομαι τώρα στους αρχηγούς των ομάδων. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα. Είχαμε πει στις 4.30. Προτείνω όμως να αρχίσουμε από τώρα. Εντάξει. Α, σε πέντε λεπτά. Καλά. Σε πέντε λεπτά προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο. Όχι, τίποτα άλλο τότε διάλειμμα 5 λεπτών μέχρι να βρει την κάρτα του και ο Σαλβαδόρ. Bien, mes chers collègues, tout le monde... Λοιπόν, έχετε όλη την κατά ψηφοφορία σας αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ. Alors, je vous propose de commencer... Προτείνω να ξεκινήσουμε ψηφίζοντας την έκθεση Torvalds για το ITER. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας, έτσι. Η Αν να αντικαθιστά τον κύριο Torvalds, αν έχετε ερωτήσει. Λοιπόν, άρθρο 2. Υπάρχει μία τροπολογία 7 του εισηγητή με μία προφορική τροπολογία που έχετε μπροστά σας. cost, overruns κλπ. deems as appropriate. Qui pour? Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές. Δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται. Το απολογεί 8 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Εννέα του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ένα κατά, εγκρίνεται. Έντεκα. οι πολλών συναδέλφων από το ΕΛΚ. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. κανεί Αποχές. Δεκτή. Ομόφωνα. Αιτιολογική σκέψη Ένα. Νέο. Του εισηγητή. Να ψηφίσουμε τις 1, 2, 3 μαζί. Όχι. Ωραία. Ένα υπέρ. Κατά. Πράσινη. Αποχή. Μία. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά. Κανείς. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία που είναι ταυτόσιμη με την δέκα υπέρ. Α, δεν είναι ταυτόσιμη, συμβατή είναι. Συγγνώμη. Ευχαριστώ τη φανή. 3 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 συμβατών υπέρ κατά η πράσινη αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του εισηγητού με έτοιμα κατά τμήματα, κατά τμήματα ψηφοφορίες το over and above the MFF ceilings μετά από έτοιμα των πρασίνων υπέρ κατά ένας. Αποχές. Δεκτή. Το υπόλοιπο της τροπολογίας υπέρ. Κατά. Πράσινη και γκουε. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε και έξι του εισηγητή μαζί. Όχι. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έξι υπέρ. Κατά. Η πράσινη. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την τελική ψηφοφορία άρχεται. Με την κάρτα μέσα στη, στη θηκούλα της. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι. 29 κάρτες, 29 ψηφίσαντες, 22, 26 υπέρ, 2 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή και στην κυρία Γέντσεν που τον εκπροσωπεί. Κατόπιν, έκθεση Βέτμαν, Ατζίλε το λένε, Ατζίλε, Ιταλία. Ή το μία και δύο μαζί μπορούμε. Όχι, δεν το θέλει η συγγήτρια. Το ένα από τους σοσιαλιστές. Τι θέλει. ΕΜ αγαπά την έκθεση αυτή ο εισηγητής. Υπέρ, κατά. Αποχές. Δεκτή. Τοπολογία 2. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. ενδιαφέρον. Γκουε και συντηρητική. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 και 4 μαζί. 3 και 4 μαζί. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Είδατε την προφορική τροπολογία του της ηγήτριας, καλωσορίζει τη συνεισφορά κλπ. Children, elderly or disabled persons to take care of these persons, to allow the workers participating in the program to reconcile trainings, etc. Ποιοι είναι Κατά. Ένας. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 από τους σοσιαλιστές. Η συγκίτρια είναι υπέρ υπέρ, κατά, ένας, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Με αντίθετη την συγκίτρια υπέρ, κατά, πλάκα έχει. 6. Η ίδια μειοψηφία, που δεν είναι ωστόσο παρελκύουσα μειοψηφία. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Για την έκθεση Βέρτμαν. 32 γίναμε, ψηφίσαμε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, 30 υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια, κυρία Βέρτμαν. Μετά, Έκθεση Νταρντέν. Όστρια Ταμπάκ. Έχουμε πέντε τροπολογίες των ιδίων συντακτών. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Μου λένε ότι η τροπολογία 3 δεν ψηφίζεται γιατί καλύπτει την παράγραφο 5. Αυτό νομίζει ο εισηγητής. Αν θέλουμε δηλαδή να μην ψηφίσουμε την τρία, δεν την ψηφίζουμε. Να ψηφίσουμε τι τροπολογίες 2, 4, 5 και 6 μαζί. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Δύο. Οποχές. Εγκρίνεται. Επτά των φιλελεύθερων. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν είναι σαφής η εικόνα. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ 14 κατά 2 αποχές εγκρίνεται. 8 και 9 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 και 11 μαζί. Ε, η συγητής είναι κατά. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Η αιτιολογική σκέψη περιλαμβάνει τη, την, ε, την επιτροπολογία 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 34 γίναμε. Αν καθυστερούμε θα φτάσουμε τους 80 τελικά. Πέρας ψηφοφορίας, 28 υπέρ 4, 4 κατά 2 αποχές. Εγκρίνεται. Alors, nous en venons au rapport... Και φτάνουμε στην έκθεση του κυρίου Ντέρεκ Βον. Le Fonds d'aide Ταμείο ενίσχυσης των απόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το κατάλογο. 28 του Ρικέ υπέρ και ο εισηγητής υπέρ είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 του Τζοβάνι Λαβία και ο εισηγητής υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπέρ 30 σοσιαλιστών εισηγητής υπέρ ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται η 31 της Γκου εισηγητής κατά ψηφιπέ τρεις 3 κατά οι υπόλοιποι σχεδόν όλοι απορρίπτεται και αποχές 32 Βέρτμαν εισηγητής κατά ψηφιπέ κατά πολύ αποχές απορρίπτεται. Ε, 33 είναι της ιδίας, αλλά εδώ είναι ο εισηγητής υπέρ, ψήφι Κατά, ένας, αποχές εγκρίνεται. 34 σοσιαλιστών, εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 35 έχει αποσυρθεί κύριε Κλούτε. 36 κότινι και Νταρντέν εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Αυτοί οι όλοι και όλοι, κατά. Αποχές, σοσιαλιστές, χάσανε. Απορρίπτεται. 37. Καταπίπτει εφόσον εγκριθεί 33, την εγκρίναμε την 33, οπότε καταπίπτει. Άρα, τώρα, εδώ έχουμε ένα συμβιβασμό α κεφαλαίο βλέπετε το κείμενο δίπλα ότι δεν θα μειωθεί σε πραγματικούς όρους το ποσό σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα ε, για την επιστημιστική βοήθεια. Ε, αυτό είναι μια, ένας μικρός επιβενιγμός για το PDP υπέρ κατά το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν περνάμε μέσω στην τροπολογία υπαριθμών 45. Α, όχι. Έχει αποσυρθεί. 46. Κοσλόφσκι, εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47. Σοσιαλιστών, εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48. Πατράου Νέβες. Είναι της κυρίας Πατράου Νέβες. Έχουμε και εξωτικέ χώρε στην Ένωση. Ονόματα είναι αυτά. Λοιπόν, σε τρία τμήματα. Το πρώτο, το, πρόγραμμα, αυτό ψηφίζουμε. Ποιο είναι υπέρ του προγράμματος, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, που δεν θα πρέπει να είναι σε ανταγωνισμό με άλλα προγράμματα στον ίδιο τομέα, κλάδο και τα οποία κατά είναι ο ο οποίος κατάλαβε, είπε η πράσινη. Ο Ρίτσαρτ και εσείς. Κατά. Αποχές απορρίψετε. Το τρίτο τμήμα. Έχει νόημα τώρα το τρίτο τμήμα. Παρόλο που το δεύτερο καταψηφίστηκε θα πρέπει να συνοδεύει άλλα μέτρα κτλ. Συγητής είναι υπέρ, Λίπερ, υπέρ, κατά. Ο κ. Μοργκάντη εποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, η τροπολογία 49 του κυρίου Κουσλόφσκη, συγητής υπέρ, άλλη υπέρ, κατά. Απόχες, εγκρίνεται. Η 50, Ρικέ, η είναι υπέρ, ψηφιπέρ, κατά. Δύο εποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα το εισηγητή που καλύπτεται από την 50, οπότε καταπίπτει. 51 ε, της γκουα εισηγητής, περιέργως υπέρ. Ασυνήθιστα υπέρ είναι. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 52 του κυρίου Κοσλόφσκη εισηγητής υπέρ. Άλλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 πίπτη γιατί εγκρίναμε την 33 η 54 της κυρίας Στροτμάν εισηγητής υπέρ ψήφι κατά κανείς αποχές εγκρίνεται 55 Κοσλόφσκι εισηγητής υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 56 της κυρίας Τροτμάν εισηγητής υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 5 και οι 58 ταυτίζονται. Έτσι δεν είναι φανή. Ε, υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με τρεις ψήφους ε, κατά. Η 57 έχει αποσυρθεί. Αφήστε δε που καταπίπτει, εν πάση 60 του κυρίου Ρικέ. Ο ΣΥΤΙΣ υπέρ. Ψηφί υπέρ. Κατά. «61» καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε 60 μαζί με την προφορική. Ναι, γιατί η προφορική ήθελε να διαγράψει μια λέξη μια τροπολογία η οποία όμως καταπίπτει. 0 επί 0, 0. Πάει 61, δεν υπάρχει. Η τροπολογία που 6 επίση καταπίπτει, 59 αποσύρθηκε, 62 επίση καταπίπτει. Τι κατόμβη τροπολογιών έχουμε εδώ. Έχουμε τώρα τρεις ταυτόσημες, 7, 64 και 65. Ψήφι Τα Κατά. Τέσσερι. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 αποσύρθηκε, 66-67 ε, γιατί είναι υπέρ, αλλά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 68, κοτεινή ταρδένη, συγητής υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, 8, του εισηγητή ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 70 καταπίπτει η 69 επίσης μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις τρεις επόμενες 71, 72, 72 όχι κρίμα 71 υπέρ Μπερές Δαρδέν νοσηγητής υπέρ ψήφι υπέρ κατά αποχές. Έχουμε μια εχθρική πλειοψηφία. 72 κοτεινή ταρτένη ηγητής υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 73 των ιδίων υπέρ και ο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι δύο επόμενες έχουν αποσυρθεί. Ερχόμαστε στην 9 και την 76 μαζί ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Από πλειοψηφία δεξιά έχουμε για τις τροπολογίες αυτές. 77 ε, και 78 έχουν αποσυρθεί. 79 Κοσλόφσκι, ο συγητής είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. 4. Αποχές εγκρίνεται. 80 έχει αποσυρθεί. 81. Μπερές Νταρντέν. υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. La majorité de droite est donc rejetée. Δεξιά πλειοψηφία απορρίπτεται. Στη συνέχεια, σε τελογικέ σκέψει. 10. Κοτεινή Νταρδένη ηγητή υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ τίποτα. Αποχή θα ψηφίσετε. Ο εισηγητής υπερψήφισε. Α, και το ΕΛΚ μαζί. Πάρα πολύ διακριτικά όμω. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε διακριτικό πλήν ισχύει. Εγκρίνεται. 13. Ε, Της Περβάς Μπερές και του κυρίου Νταρτέ, εισηγητής υπέρ, ψήφι κατά, απόχες, εγκρίνεται. 12. Γκούε, εισηγητής υπέρ, ψήφι κατά, απόχες, εγκρίνεται. Η 11 κατέπεσε. 14 και 15 μαζί. Εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. 16 Μπέρες Δαρντέν. Εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. 2 κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 καταπίπτει. 18 Ρικέ, εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά τρεις, τέσσερις αποχές εγκρίνεται. Η 19 καταπίπτει όπως και η 20 που έχει αποσυρθεί και 21 καλύπτεται. 21 μου λέγουν ότι καταπίπτει, παρόλο που δεν το γράφει. Η τροπολογία 1 του εισηγητή καταπίπτει. Η τροπολογία 2 του εισηγητή θα πρέπει να ψηφιστεί ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 22 καταπίπτει. 23. Κοτινή Νταρντέν Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 Μπέρες Νταρντέν Συγητής υπέρ, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 25-26, Νταρτέν Κοτινή. Από έχουν υποβάλει την ίδια τροπολογία, αλλά όχι μαζί αυτή τη φορά. Τένις παίζουν, πότε μόνοι τους, πότε διπλό. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 του Ρικέ, ο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο, παρακαλώ. Πέρασε. Όσο πάει η ώρα πληθαίνουμε. Ξυπνήσαν από τη σιέστα. Πέρασε. Α, η Αγγέλικα μόλις έφτασε και ψήφισε. 37 Δεν ξέρουμε τι ψηφίζει η Αγγέλικα. Α, ξέρουν. Δεν είναι δημόσια ψηφοφορία, δεν μυστική είναι. 33 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Alors, euh, Έχουμε κάτι μεταφορές να ψηφίσουμε. Τζοβάνι, Λαβία. Έχεις μια μεταφορά πιστώσεων εδώ. Προϋπολογισμός 2013, τμήμα 3, Επιτροπή. Αντιστοιχούν στα δύο προγράμματα προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Προτείνω να ψηφίσουμε μπλοκ. No. Ça me fait fumer. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε πρώτα το Ατζίλε, Ιταλία. Ποιος είναι υπέρ. Κα, υπέρ είπα, υπέρ, κατά. Αποχές. Ωραία. Δεύτερον, Αύστρια Ταμπάκ, Εντάξει, τα μπακ λέει, αλλά δεν είναι για να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση καπνού, να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνουμε. Πράγμα που συμβαδίζει και με αυτά που ψηφίσαμε πριν. Μήπως κάμια άλλη μεταφορά δεν έχει άλλο θέμα στην σε διάταξη. Όχι, λύεται η συνεδρία σας. Κατευχαριστώ.